Good uh, afternoon, early evening. Καλησπέρα σας. Καθίστε παρακαλώ. I would like to uh, welcome all uh, representatives of the Θέλω να καλωσορίσω όλους τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων καθώς και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να καλωσορίσω και τον Νταμίρ Ματερλιάν στα δεξιά μου, στα αριστερά μου για σας, τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Κρατικό Κοινοβούλιο. Θα συμπροεδρεύσει αυτή την ανταλλαγή απόψεων και μεταξύ άλλων θα ολοκληρώσουμε την διακοινωνιστική μας συνάντηση σήμερα. Επίσης, θέλω να καλωσορίσω του προσώπου από το Κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου που είναι παρόντε για την ανταλλαγή απόψεων. Όπω ε, ξέρετε, σήμερα θέλουμε να συζητήσουμε πώς θα έχουμε έναν ευρωπαϊκό προπολογισμό για το επόμενο πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο κατάλληλο να αντιμετωπίσει τι παγκόσμιες προκλήσει που αντιμετωπίζουμε. Είναι ένα ιδιαίτερα επίκαιρο θέμα, όπω γνωρίζετε όλοι, εκτός ε, και αν ήσασταν στον Άρη τις τελευταίες μέρες ή εβδομάδες. Είναι λοιπόν ένα ιδιαίτερα επίκαιρο ζήτημα ο πρόεδρος του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισελ, δημοσίευσε μία νέα εκδοχή της πρότασης του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου την Παρασκευή και μία ειδική συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα λάβει χώρα την επόμενη Πέμπτη σε δύο ημέρες για το πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο και τα συναφή ζητήματα. Η σημερινή μας συζήτηση λοιπόν λαμβάνει χώρα έναντι ενό φόντου εντόνων διαθεσμικών συζητήσεων. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερη η χρονική συγκυρία για την ανταλλαγή αυτή απόψεων. Να ξεκινήσω υπενθυμίζοντας ότι κατά τη διάρκεια των ε, ευρωπαϊκών εκλογών ε, πέρσι οι πολίτες κάλεσαν την Ένωση να, να λάβει δράση για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και ο κόσμος. Δεν πρέπει να τους απογοητεύσουμε αναμένουν από την Ευρώπη να καταπολεμήσει την κλιματική αλλαγή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη νέα πράσινη συμφωνία και τον μηχανισμό δίκαιης μετάβαση προκειμένου η Ευρώπη να γίνει η πρώτη ουδέτερη κλιματικά οικονομία μέχρι το 2050. όμω την πρόταση που βρίσκεται τώρα επιτάπητο, τα κονδύλια για τη χρηματοδότηση αυτού του κόστου στόχου αφαιρούνται από άλλα σημαντικά προγράμματα όπω το Horizon Ευρώπη, η Γεωργία και το Erasmus+. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν μπορούμε να το δεκτούμε. Δεν ε, μπορείς να ξεγυμνώσεις τον Πίτερ για να ντύσεις τον Πολ και άλλες ε, ε, προκλήσεις είναι η ψηφιακή επανάσταση, η ανεργία, μεταναστευτικές πιέσεις, γεωπολιτική αστάθεια. Ωστόσο, τα χρηματικά στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί μέχρι τώρα και πάλι στην πρόταση του Μισελ, ε, είναι μεγάλη απογοήτευση για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η πρόταση είναι πολύ πιο κάτω από όσα είναι απαραίτητα και οι πολίτες αξίζουν ένα ρεαλιστικό προϋπολογισμό για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που ανέφερα και πολλές άλλες. Να τονίσω απλώ ότι στη σημερινή πρόταση το συνολικό επίπεδο ω ποσοστό του καθαριστού εγχωρίου εισοδήματο του επόμενου δημοσιονομικού πλαισίου θα είναι ουσιαστικά χαμηλότερο από το σημερινό για 27 κρατημέλη Παρόλε τι πρόσθετε ευθύνε, τι φιλοδοξίε και τα 7 έτη οικονομικής ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, ο τρόπο που ο Ευρωπαϊκό Προπολογισμό χρηματοδοτείται θα πρέπει να εξυγχρονιστεί. Μέχρι τώρα το σύστημα Ευρωπαϊκή Ένωση Ιδίων Πόρων αποκλειστικά σχεδόν βασίζεται στι εθνικέ συνεισφορέ ει ε, βάρο του εθνικού εισοδήματο. Υπάρχουν δυνατότητε να έχουμε μια επικοδομητική μεταρρύθμιση. Να τονίσω ότι οι προτινόμενες αλλαγές στην πρόταση του Σάρλ Μισελ είναι ένα άνοιγμα προ αυτή την κατεύθυνση. Για πρώτη φορά, σε πάνω από 40 χρόνια, νέε κατηγορίε ιδίων πόρων θα Ωστόσο, αυτή τη στιγμή μιλάμε περισσότερο για μια συμβολική κίνηση παρά για μια πραγματική αλλαγή. Η κατάργηση των επιστροφών επίσης θα πρέπει να εξασφαλιστεί για να διασφαλίσουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και δικαιοσύνη. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι αυτός ε, είναι, αυτή είναι ήδη η πόρη, δεν είναι ευρωπαϊκή φόρη. Το σύστημα η λοιπόν θα συνεχίσει να βασίζεται σε μια νομικά δεσμευτική συμφωνία ε, με τα κράτη-μέλη και θα βασίζεται στην απόφαση των δύο πόρων που κυρώνεται από τα Εθνικά Κοινοβούλια που θα συνεχίσουν να έχουν την κυριαρχία στα φορολογικά. Όμως στην Ευρώπη πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά ε, απέναντι στις άλλες μεγάλες δυνάμεις. Η Ευρώπη νομίζω μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία μόχλευσης για τις εθνικές οικονομίες ε, για να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις, να προωθήσουν την ανταγωνιστικότητα και την αριστεία σε τομείς όπως η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οδηγούν στα καλύτερα αποτελέσματα. Υπάρχει κάτι σαν οικονομίες κλίμακας για κάποιες δραστηριότητες και κάποιες συναλλαγές όπου Όντω, το να έχει κανεί μεγάλο μέγεθο αποτελεί πλεονέκτημα. Η Ευρώπη δεν αντικαθιστά δεν ούτε υποκαθιστά την Εθνική Κοινοβούλια και την εθνική του κυριαρχία. Ο προπολογισμό τη Ευρώπη είναι επίση ένα προπολογισμό επενδύσεων. Όλε οι χώρε υποφελούνται από τι προστιθέμενη αξία αυτού του ευρωπαϊκού προπολογισμού, ακόμη και οι καθαροί συνεισφέροντε. Προσπαθώντα βραχυπρόθεσμα να ξεκονομήσουν χρήματα, τα κράτη-μέλη κινδυνεύουν να ε, θέσουν σε κίνδυνο τι ευρωπαϊκέ αξίε μέσω πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Ξέρω ότι οι απόψεις που ακούστηκαν στη διάρκεια του Συμβουλίου δεν είναι απαραίτητα οι απόψει ε, των βουλευτών των Εθνικών Κοινοβουλίων. Γι' αυτό ανυπομονώ να κάνουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων μαζί σα, ε, καθώ εσεί εκπροσωπείτε του πολίτε ε, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για το πώ μπορούμε να κάνουμε τον προπολογισμό κατάλληλο για να βοηθήσουμε την ευρωπαϊκή και τι εθνικέ οικονομίε να αντιμετωπίσουν τι πολλέ παγκόσμιε προκλήσει που επίκυνται. πριν να ξεκινήσουμε τις συζητήσεις, να σας ε, πω ποιοι είναι οι κανόνες οργάνωσης της συζήτησης που θα πρέπει να σεβαστούμε. Διαφορετικά δεν θα μας φτάσει ο χρόνος. Λοιπόν, για να ζητήσετε το λόγο. Καταρχήν, να τονίσω ότι ο συνήθως θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι θα μπορέσουν ε, να τοποθετηθούν όσο δυνατόν περισσότεροι συμμετέχοντες. Καθώ έχουμε μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων, σας παρακαλώ να κατανοήσετε ότι μετά από τις παρουσιάσει του πάνελ, που θα προσπαθήσουμε επίση να τηρήσουμε εντό κάποιων χρονικών ορίων, πιθανότατα δεν θα είναι δυνατό σήμερα όλοι να πάρουν το λόγο. Και γι' αυτό σας ζητώ ευγενικά να περιοριστείτε στα δύο λεπτά στις παρεμβάσεις σας και θα βλέπετε και το ρολόι στην οθόνη. Ανάλογα με την εξέλιξη των συζητήσεων μπορεί να χρειαστεί να αλλάξουμε αυτό το χρονικό όριο. Θα βρείτε ε, μπροστά σας ε, κάποιες κάρτες αγόρευσης. Με αυτές μπορείτε να ζητήσετε το λόγο. Αν ε, θέλετε να πάρετε το λόγο, παρακαλώ συμπληρώστε τις κάρτες αυτές και δώστε τις στους κλητήρες στην αίθουσα. Αυτό ισχύει και για τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων. Γενικά θα προσπαθήσουμε να διαιρέσουμε το χρόνο αγόρευσης σύμφωνα με την ακόλουθη φόρμουλα. Δύο βουλευτές από τα Εθνικά Κοινοβούλια και θα ακολουθεί ένας Ευρωβουλευτής. Λοιπόν, κατόπιν όλων αυτών θα δώσω τώρα το λόγο με τα χαράς στον κύριο Ματέλια για να συνεχίσει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην αρχή αυτής της συνεδρίασης έχουμε αξιομιλητές. Ο πρώτος είναι ο κύριος Γιάνν Όλμπριχτ, ο οποίος ε, είναι συνεισηγητής για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Έχετε το λόγο κύριε Όλμπρικτ, αλλά μόνο για πέντε λεπτά παρακαλώ. Πέντε λεπτά σε κοινοβουλευτικού όρου δεν είναι άσχημα. Σα ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μοιραστώ μαζί σα και με του συναδέλφου από τα Εθνικά Κοινοβούλια τι εργασίε μα. Και να σα υπενθυμίσω ότι όλο το πακέτο για το πολιτιστικο δημοσιονομικό πλαίσιο περιλαμβάνει διάφορα στοιχεία και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό να το κατανοήσουμε, ότι όλη η συζήτηση δεν έχει να κάνει με ένα μόνο στοιχείο, αφορά όλα τα στοιχεία που εμπεριέχονται. Και αυτό που μόλι επισημένα ο πρόεδρο. Ο κανονισμό για το πολιτιστικο δημοσιονομικό πλαίσιο, για το πόσα χρήματα θα μπουν στον προπολογισμό, ποια θα είναι τα βασικά στοιχεία, οι βασικέ πολιτικέ που θα χρηματοδοτηθούν, τι θα γίνει με το οικοδόμημα του προπολογισμού και του εσωτερικούς μηχανισμούς, αλλά και πώς θα λειτουργήσει ο προϋπολογισμός. Αυτό, αφανώς. Κατά δεύτερον, ήδη μπορεί το εξήγησαν οι συνάδελφοι, νομίζω ότι είναι σαφές. Το τρίτο. Πάνω από 40 κανονισμοί, οι οποίοι σχετίζονται με τις μεταφορές από την Παταμία Συνοχής, από τον ορίζοντα κτλ. Που πλέον έχουν αναλάβει οι ε, στο Κοινοβούλιο. Και το τέταρτο θέμα είναι το κράτο δικαίου. Άρα, καταρχά, έχουμε βάσει τη απόφαση ε, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μια ομόφωνη απόφαση που προποθέτει προϋποθέτει τη συγκατάθεση του Κοινοβουλίου. Στο δεύτερο στοιχείο έχουμε μια διαφορά και το εξήγησε ο συνάδελφο για του ίδιου πόρου. Είναι διαφορετική διαδικασία και ο οι κανονισμοί για τι διάφορε πολιτικέ αποφασίζονται βάσει συναπόφαση. Εδώ λοιπόν έχει ισχυρό ρόλο να παίξει το Κοινοβούλιο μέσω των διαπραγματεύσεων. Και το τέταρτο στοιχείο αφορά το νέο κανονισμό για το κράτο δικαίου, όπω προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε ό,τι αφορά το πρώτο στοιχείο τώρα, γιατί είμαι συνεισηγητή ε, στο πρώτο θέμα σε ό,τι αφορά το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Στην προηγούμενη θητεία παρουσιάστηκε η άποψη του Κοινοβουλίου για το ποιο θα πρέπει να είναι το ποσό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη και το Brexit, λαμβάνοντας υπόψη και τις νέες προτεραιότητες. Και υπό τον ε, όρο ότι θέλουμε να έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση στο ίδιο επίπεδο. Στο ίδιο επίπεδο δηλαδή χωρίς τη Μεγάλη Βρετανία. Αν θέλουμε να διατηρηθεί στο ίδιο επίπεδο η Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς τους Βρετανούς, είναι σαφές ότι υπάρχει ένα ε, δημοσιονομικό κενό. Αυτό το κενό λοιπόν κάπως πρέπει να το καλύψουμε. Αν θέλουμε λοιπόν η Ευρώπη να παραμείνει επαναλαμβάνω στο ίδιο επίπεδο. Είτε λοιπόν αυτό το κενό θα καλυφθεί από μεγαλύτερε εθνικέ συνεισφορέ ή από ίδιου πόρου, είτε από περικοπέ στι πολιτικέ. Αυτό λοιπόν που κάνουμε τώρα είναι μια πραγματική, επί τη ουσία, πολιτική συζήτηση για το τι θέλουμε τελικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να παραμείνει στο ίδιο επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστούμε πιο πολλά χρήματα λόγω του Brexit ή θέλουμε μήπως να περιοριστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόταση που λάβαμε και την οποία περιέγραψε ο πρόεδρο, καταδεικνύει ότι ο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά τι διμερεί συναντήσει, γιατί δεν ήταν δική του ιδέα αυτή, ήταν αποτέλεσμα και απορία των δημερών συναντήσεων για εξέβρεση ε, και ομοφωνιάς. Η πρόταση λοιπόν τι συνεπάγεται ότι θα περιοριστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, το επίπεδο φιλοδοξίας, το πεδίο εφαρμογής και δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Γι' αυτό λοιπόν η άποψη των διαπραγματευτών για το πολιτισμικό πλαίσιο είναι ότι θα το απορρίψουμε αυτό ως πρόταση. Γιατί πιστεύουμε ότι η προσέγγιση αυτή ουσιαστικά περιορίζει τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό μπορούμε να το δείξουμε σε διάφορα προγράμματα. Γιατί ο πιο περιορισμένος προπολογισμό σημαίνει λιγότερες δαπάνες σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα προγράμματα. Κοιτώντας τα, την πρόταση του Προέδρου της Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δεν είναι γενικόλογη, αφορά συγκεκριμένε περικοπέ συγκεκριμένε πολιτικέ, ε, ό,τι αφορά την πολιτική άμυνα 50%. Ε, έρευνα, κοινωνικά, συνανοχή. Παντού προβλέπονται συγκεκριμένε περικοπέ. Γι' αυτό λοιπόν η δική μα θέση σήμερα είναι σαφή αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε στο Κοινοβούλιο είναι μια συνεργασία με όλους τους συζητητέ. να υπάρχει μια συνοχή σε ό,τι αφορά την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε ό,τι αφορά όλες τις πολιτικές ομάδες και ως τώρα υπάρχει αυτή η συνοχή, θα προασπιστούμε τι φιλοδοξίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το πεδίο εφαρμογή, τι ενέργειε, τι δράσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν στην παρούσα φάση των διαπραγματεύσεων η απάντησή μα είναι όχι. Ευχαριστούμε κυρία Ολμπρέχτ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση αυτή και σας ευχαριστώ που σεβαστήκατε και το χρονικό όριο. Δεύτερος τώρα ο μιλητής είναι η κυρία Μαργαρίτα Μάρκες. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, θα μιλήσω πορτογαλικά. Στο <laughs> ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν ε, θέλω να αναφερθώ στη σημασία αυτού του είδους των συνεδριάσεων και να ανταλλάξουμε απόψεις μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών βουλευτών. Ήδη όπως είπαμε και στην Ολομέλεια, είχα την ευκαιρία να είμαι και από την άλλη πλευρά, να βρίσκομαι εδώ, αλλά εκπροσωπώντας το Πορτογαλικό Κοινοβούλιο. Και αυτή η συνεργασία είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι πολύ σημαντική στη συζήτηση για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε από αυτά που υπόθηκαν από τον ε, συνεισηγητή, τον κύριο Όλμπριχτ, η κατάσταση είναι εύκολη. Θα έλεγα μάλιστα ότι είναι δύσκολη. Όμως είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε και να ακούσουμε τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί το τελευταίο πράγμα που θέλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι να βρεθεί στη μέση μιας διαθεσμικής κρίσης, μιας διοργανικής κρίσης. Εμείς βρισκόμαστε τώρα στην αρχή του νέου θεσμικού κύκλου με νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, νέο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτός ο θεσμικός κύκλος έχει μια θεμελιώδη πρόκληση να αντιμετωπίσει. Είναι να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η πρώτη πρόκληση. Και εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, είναι ενωμένο και ασχολείται πλήρως με αυτό. Αν είχαμε αμφιβολίες, ε, αρκούσε να διαβάσουμε την επιστολή που επέγραψαν την περασμένη εβδομάδα, από, που υπεγράφει από τους ε, τέσσερις επικεφαλείς των τεσσάρων μεγάλων πολιτικών ομάδων του Κοινοβουλίου. Γιατί εμείς τι θέλουμε καταρχήν, να απαντήσουμε στις προσδοκίες των πολιτών. Εμείς ε, έχουμε εκλεκτεί από τους Ευρωπαίους πολίτες σε μας κατέθεσαν ε, μία σειρά προσδοκιών ε, και όλοι μας αντιλαμβανόμαστε ποια ήταν τα θεμελιώδη σημεία, ποιες ήταν οι προσδοκίες των πολιτών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παραδείγματο χάρη, η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής ήταν ένα ε, θέμα που κυριάρχησε στις προεκλογικές εκστρατείες όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, αλλά μια δίκαιη μετάβαση που να μην αφήσει κανέναν πίσω, που να μην προκαλέσει νέες ανισότητες. Ήταν επίσης ένα θέμα που ήταν ε, στα εκλογικά θεματολόγια σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, πρόθεση της στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη σύγκληση και τη συνοχή, η κινητοποίηση των νέων για την συμμετοχή στην πολιτική, για καλύτερη γνώση τη Ευρώπη. Όλα αυτά είναι στο πολιτικό μα θεματολόγιο και γι' αυτό εμεί έχουμε τη φιλοδοξία αυτή σε σχέση με τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, γι' αυτό εμείς λέμε ότι αυτός ο προπολογισμό που είναι τώρα επιτάπητος δεν αρκεί. Γιατί εμείς ε, τι ε, πιστεύουμε, τι ακούσαμε, όλοι οι ηγέτες των κρατών μελών, τα μέλη της Κομισιόν, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όταν μιλάνε για τις προτεραιότητες για τις φιλοδοξίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση, φαίνεται να συμφωνούν με τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όμως, στη συνέχεια, όταν αυτές τις προτεραιότητες τις μετατρέπουν ε, σε κονδύλια, ε, τότε βλέπουμε ότι βρίσκονται πάρα πολύ μακριά από την ικανότητα να μπορούν να καλυφθούν αυτές οι προτεραιότητες. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι με αυτόν τον προπολογισμό εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε την συγκατάθεσή μας εμείς ε, ακόμη και αν ε, ε, σε αυτή τη φάση είναι απαραίτητο, θέλουμε μεγαλύτερη άμεση συμμετοχή των κρατών μελών. Συνειδητοποιούμε ότι εξακολουθεί να είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο και θα συνεχίσει στο επίπεδο αυτό να είναι απαραίτητη η συμμετοχή των κρατών μελών. Όμως γνωρίζουμε ότι ο προπολογισμό μπορεί να αυξηθεί με ίδιους πόρους, με νέους ίδιους πόρους που δεν θα ποινικοποιούν τους πολίτες, που θα σχετίζονται με στόχους πολιτικούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής, ο φόρος επί των πλαστικών, ο φόρος ε, για τις συναλλαγές ε, του άνθρακα. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με πολιτικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν όμως και άλλοι είδη οι οποίοι προκύπτουν από τα ωφέλη της εσωτερικής αγοράς. Παραδείγματος χάρη φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ή ένα άλλο παράδειγμα, φόρος επί των ψηφιακών εταιριών. Εμείς διαφορετικά δεν μπορούμε να είμαστε συναφείς. Συναφείς ως προς το εξή ότι ε, την ε, χρήση των ε, ιδίων πόρων θα την ευθυγραμμίσουμε με τους πολιτικούς στόχους. Γιατί εμείς ε, τι θέλουμε, να ψηφίσουμε και να εγκρίνουμε και να διορθώσουμε ένα πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ένα προπολογισμό που πρέπει να υφίσταται το 2021, αλλά φυσικά αυτό δεν μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε τίμημα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, you, Mrs. κυρία Μάρκες και πήρατε 35 δεύτερα από το χρονομιλία του κυρίου Όλμπριχτ. Δεν πειράζει όμω τι να κάνουμε. Και προχωράμε με τον κύριο Χώσε Μανουέλ Φερνάντε, τον επόμενο μιλητή, ο οποίο είναι συνεισηγητή για του ιδίου πόρου. Έχετε το λόγο για 5 λεπτά. Ευχαριστώ και θα μιλήσω γαλλικά. Έχουμε έναν ε, προπολογισμό περιορισμένο και με τον περιορισμένο αυτό προπολογισμό θέλουμε να τα πετύχουμε όλα. Έχουμε έναν προπολογισμό ο οποίο έχει ε, τεράστια προστιθέμενη αξία και διαρκώ επαναλαμβάνουμε και τονίζουμε ότι όλοι τα θεσμικά όργανα είναι στο, στο 7% Θέλουμε μια Ευρώπη με γεωπολιτικό βάρο που θα ανταποκριθεί στι προκλήσει ε, τις οποίες από κοινού μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ε, πιο καλά για να μην ταπανούμε πιο πολλά χρήματα ε, με κάθε κράτος μέλος που θα έπρεπε εναλλακτικά να κάνει τι δουλειές αυτέ. Μιλάμε για την παλιά πολιτική. Μιλάμε για μια πολιτική παραδοσιακή, όπως η πολιτική γεωργίας. Έχουμε νέες προκλήσεις όμως, θα πρέπει να τις ε, αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε έναν ε, προπολογισμό που 85% προέρχεται από τα κράτη-μέλη, από το ΑΕΠ και από το ΦΠΑ. Και 15% μόνο ε, είναι δικά μας, δική μας δασμή. I want my money back. Θέλω τα λεφτά μου πίσω λες και κάθε υπουργό θεωρεί ότι είναι δικά του τα χρήματα αυτά και θα πρέπει να το επιστραφούν. Να πούμε ότι η Γαλλία και η Γερμανία από κοινού έχουν 38% των δαπανών. Αυτό τι σημαίνει ότι οι δύο κράτη-μέλη ε, αντιπροσωπεύουν ε, από κοινού το 38%. Αυτό προφανώς τους δίνει ε, μια δύναμη σε ένα τέτοιο προϋπολογισμό που πρέπει να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε σε όρους καθαρών εισφορέων και καθαρών δικαιούχων. Όλος ο κόσμος ωφελείται και αυτό αποδεικνύεται από μελέτες που καταδεικνύουν ότι κάθε κράτος μέλος, ακόμα και αν δεν έπαιρνε τίποτε από τον προπολογισμό, έχει τεράστιο όφελος. Λόγω της ενιαίας αγοράς, λόγω της εσωτερικής αγοράς. Ξέρουμε όμως ότι φυσικά ε, έχουν, λαμβάνουν και πόρους και υπάρχουν και επιστροφές, επιστροφές και αποζημιώσεις από των επιστροφών. Κοιτάξτε για τι γίνεται. Εμείς καταλήξαμε σε ένα α, ποσοστό, 1,3% του ΑΕΠ. Δεν είναι μαγικός αριθμός αυτός, είναι αυτό που χρειάζεται για τη χρηματοδότηση του προπολογισμού. Με μια αρχή η οποία αρχή που μα βρίσκει σύμφωνο, ότι αυτοί που δεν πληρώνουν θα πρέπει να πληρώσουν. Δηλαδή οι ψηφιακέ εταιρείε οι μεγάλε θα πρέπει να πληρώσουν. Αυτό είναι επιτάπητο. Αυτή η πρόταση του κυρίου Μισέλα για του ιδίου πόρου είναι προ τη σωστή κατεύθυνση. Αντίθετα με την πρόταση για το πι δελτα πι. Είναι στο σωστό δρόμο γιατί μιλάει για αφορολόγηση του πλαστικού σε ό,τι αφορά το σύστημα ETS για την εμπορία ρήπων. Και να κινηθούμε σε ό,τι αφορά τους ίδιους πόρους στην επιβολή φόρων στις μεγάλες επιχειρήσεις. Επίσης, θα πρέπει να υπάρξει μια εναρμόνιση επί της αρχής αυτής σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λόγω φοροδιαφυγής και εξεβλήματος χρήματος χάνουμε 7 χρόνια προπολογισμού. Αντίστοιχο ποσό. Είναι απίστευτα τα ποσά. Και προφανώς το πρέπει να κάνουμε προσπάθειες για να αποφύγουμε επιπλέον επιβάρυνση των πολιτών. Να είμαστε επίσης, ε, να συνειδητοποιήσουμε το εξής, ότι είμαστε σε ένα κόσμο όπου είμαστε το μοναδικό κοινοβούλιο με δικαίωμα α, ε, μα, καθορισμού του προπολογισμού, αλλά όχι σε ό,τι αφορά τα έσοδα. Και τίθεται επίση το θέμα τη ομοφωνία. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι χρειάζεται επικύρωση από όλα τα εθνικά κοινοβούλια. Θα μπορέσουμε λοιπόν να συνενέσουμε σε ό,τι αφορά το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο μόνο αν υπάρχει συμφωνία για τους ίδιους πόρους. Για παράδειγμα, τα πρόστιμα. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Αποτελεί ε, ένα έσοδο σε ό,τι αφορά ε, τις πολιτικές ανταγωνισμού, αλλά προέρχονται από τον προπολογισμό. Στον επόμενο χρόνο, το έτο, έτος, ε, επιστρέφουν στι τσέπε του κάθε κρατου μέλους σε ό,τι αφορά τις εισφορέ. Κατά αναλογία δηλαδή των, προσφορών, των εισφορών του κάθε κράτου μέλους. Αυτό είναι απαράδεκτο πραγματικά. Και ένα άλλο στοιχείο είναι η απλοποίηση. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσει και τις επιστροφές έχουμε να πούμε το εξή. Σε ό,τι αφορά τα ελληνικούς δασμού. Θεωρώ ότι είναι υπερβολικό το γεγονό ότι τα κράτη-μέλη κρατούν 20% των τελών. Θεωρώ ότι 10% θα ήταν υπεραρκετό ποσοστό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Φερνάνδε. Και τώρα να δώσουμε το λόγο στην Βαλερή στην συγκεκριά, για τους ίδιους πόρους. Έχετε το λόγο. Πέντε λεπτά. Ε, Ευχαριστώ. Χαίρομαι που συμμετέχω σε αυτό το πάνελ που θα μου επιτρέψει να δείξω ότι ο ευρωπαϊκό προπολογισμό στι διάφορε συνιστώσει του και στα έσοδα και στα εξόδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ω τέτοιο και να υπηρετήσει τι ευρωπαϊκέ μα πολιτικέ και να μα επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τι παγκόσμιε προκλήσει. Αν δούμε στο παρελθόν τα διάφορα δημοσιονομικά πλαίσια, το κάθε ένα εξυπηρέτησε μια μεγάλη πολιτική, ένα στόχο από το 88 στο 93, εσωτερική αγορά 94-99, οικονομική και νομισματική ένωση 2000-2006, μεγάλη διεύρυνση 2007-2013, συνέχιση της διεύρυνσης και στρατηγική της Λισαβόνας 2014-20, βιώσιμη και φύση ανάπτυξη. Κατά την άποψή μου, το μελλοντικό πλαίσιο θα πρέπει να ε, συνοδεύσει δύο στρατηγικές ευρωπαϊκή κυριαρχία και οικολογική μετάβαση. Επί της ουσίας θα πρέπει να διασφαλίσουμε ε, μια κυριαρχία διατροφική τη δημιουργία μέσων κοινή άμυνο, ένα ε, πρόγραμμα διαστημικό που θα μα επιτρέψει να ε, αντιμετωπίσουμε τι άλλε μεγάλες δυνάμει. Σε ό,τι αφορά το κλίμα και το περιβάλλον θα πρέπει οι δαπάνε μα να έχουν ε, ένα θετικό όφελο, όχι μόνο μέσω προγραμμάτων όπω το LIFE ή το ορίζοντα, αλλά σεβόμενοι και τη Συμφωνία των Περισσίων. Αλλά δεν μετρούν μόνο οι δαπάνες και τα έσοδά μας μπορούν να απαντήσουν τις προκλήσει. προκλήσεις. Ε, Παραδείγματο χάρη, αναφέρθηκε ήδη, υποστηρίζουμε τη δημιουργία μιας εισφοράς ε, στα πλαστικά. Σημαίνει αυτό ότι τα κράτη θα πρέπει να δίνουν στον ευρωπαϊκό προπολογισμό 80 λεπτά του ευρώ. Συζητάμε ακόμα αν μιλάμε για ένα ευρώ ή για 80 λεπτά. Δεν έχει ακόμη θεσπιστεί. Ανακυλώ ε, πλαστικών που δεν έχουν ανακυκλωθεί στο σύνολο των πλαστικών ε, αποβλήτων που παραγόνται σε μια χώρα. Πρόκειται για ένα πραγματικό εργαλείο ε, που χρησιμοποιεί η Κομισιόν στη στρατηγική της κατά των πλαστικών και να προστατεύσει τους ωκεανούς και το περιβάλλον και συμμετέχει ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός. Επίσης, υποστηρίζουμε την ολοκλήρωση του συστήματος των εσόδων από το σύστημα ανταλλαγής ποσοστώσεων των εκπομπών του άνθρακα. Αυτός ο μηχανισμός ε, θα πρέπει πρώτη πρώτη του 2021 να έχει τεθεί σε εφαρμογή το νωρίτερο ε, για να μπορέσουν να σεβαστούν και τους κανόνες μας οι τρίτες χώρες. Ε, έτσι λοιπόν θα επιτρέψουμε να αποφύγουμε και τη διαρροή άνθρακα ε, που οδηγούν στη μεταγκατάσταση των επιχειρήσεών μας επειδή έχουμε ε, πολύ υψηλού κανόνες σε ό,τι αφορά τη ρήπανση. Υπάρχουν και, άλλες, άλλοι πόροι που αναφέρθηκαν παρνούντος χάρη προκειμένου να υπάρχει δίκαιη φορολόγηση των πρωταγωνιστών που ωφελούνται από την Ευρωπαϊκή αγορά. Όμως στην Ευρώπη έχουμε αυτή την κουλτούρα της συνεισφοράς στην ευημερία της κοινωνίας και αυτό περνά απαραίτητα ε, από ε, αυτά τα μέτρα για να ενισχύσουμε την ισότητα. Θα σταματήσω εδώ, απλώς θέλω να πω δύο λόγια για να αντιδράσω στο διαπραγματευτικό κουτί που παρουσιάστηκε από το Σόρι Μισελ την περασμένη εβδομάδα. Ε, σίγουρα θα συμφωνήσω με το Ζωζέ Μανουέλ και μάλιστα θα πάω και πιο πέρα. Ναι, οδεύουμε προ την κατεύθυνση. Πραγματικά είναι ότι ο Σέλ Μισελ έκανε πολύ μεγάλη δουλειά, εξέτασε τι θέσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αυτό είναι σημαντικά. Υπάρχουν ε, θετικά μηνύματα, όμω ε, δεν ε, τα έχουμε βρει ακόμη, ούτε για του ίδιου πόρου. Γιατί αν ξύσουμε λίγο, θα δούμε από κάτω ότι θα πρέπει να είμαστε σόφρονε ό,τι αφορά τη συνεισφορά των πλαστικών. Θα σας υπενθυμίσω το πλαίσιο. Εδώ και χρόνια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά νέους ίδιους πόρους. Επίσης, εδώ και χρόνια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά την κατάργηση των επιστροφών. Και σήμερα, στην πρόταση, έτσι όπως παρουσιάστηκε την Παρασκευή, έχουμε νέους πόρους, ναι, τη συνεισφορά πλαστικών, αλλά με επιστροφή. Δηλαδή αυτό έρχεται να σαμποτάρει την ίδια την αρχή, ε, γιατί δεν υπάρχει πλέον στο κίνητρο στο πνεύμα αυτού του ιδιοπόρου. Έχουμε πραγματικό πρόβλημα λοιπόν. Το δεύτερο θέμα, ο Ζωζέ το είπε, γίνεται επίκληση στο να εισάγουμε νέους πόρους στο ε, δημοσιονομικό πλαίσιο, όμω είναι πολύ αόριστη διατύπωση και δεν αρκεί. Θα πρέπει να έχουμε πραγματική σαφή δέσμευση από την πλευρά των κρατών μελών για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο σε σχέση με την εισαγωγή νέων ίδιων πόρων. Γιατί αν αυτό δεν λέγεται ξεκάθαρα και δεσμευτικά, σίγουρα για 20 χρόνια δεν θα έχουμε καμία μεταρρύθμιση. Θα σταματήσω εδώ και ελπίζω να σας έδειξα ότι θα πρέπει ο μελλοντικό προπολογισμό Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι ένα εργαλείο που θα εξυπηρετεί την κυριαρχία. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Χαγιάν. Θα μείνουμε στα γαλλικά και θα περάσουμε τώρα το, σε δύο αμβουλευτές από την Γαλλία, τον κύριο Βινσάν Μπλε. Α, όχι, στον κύριο Ζαν ε, Φρανσουά από την ε, Ουλευτική Επιτροπή Οικονομικών ε, Θεμάτων της Γερουσίας της Γαλλίας. Οπότε έχετε το λόγο, παρακαλώ. You can say better <laughs> Okay. <laughs> mesdames et messieurs. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, αγαπητοί συνάδελφοι. Το επόμενο πολιτιστικό πλαίσιο θα καθορίσει του στόχου και τι φιλοδοξίε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2027. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγορείται για δράνεια και είναι η πηγή κάθε κακού, υποτίθεται. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τι θα γίνει στο μέλλον. Θα χρειάζομαστε και έχουμε μια ευθύνη συλλογική για να επιτρέψουμε, να μπορέσουμε να βρούμε μια απάντηση. Και θα πρέπει να ακουστούν και τα εθνικά κοινοβούλια εδώ από την αρχή των διαπραγματεύσεων. Η γερουσία της Γαλλίας έχει εγκρίνει διάφορες ε, ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να επισημοποιήσουμε τη θέση μας ό,τι αφορά το επόμενο πολιτές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά και την επερχόμενη σύνοδο για το θέμα αυτό. Αυτός ε, ο προπολογισμό ε, είναι 1,11 του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η πρόταση όμως ε, προκαλεί μεγάλες διαφωνίες μεταξύ των πολιτικών ομάδων και κομμάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλάει για νέες προτεραιότητες έρευνα, ασφάλεια, έλεγχο των συνόρων και εράσμος και η Γαλλία συμφωνεί σε ό,τι αφορά τι προτεραιότητε αυτέ για να ανταποκριθούμε στι προκλήσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει περικοπή στι παραδοσιακέ πολιτικέ, όπω η πολιτική γεωργία, η πολιτική συνοχή. Και εδώ βλέπουμε 15% και 10% αντίστοιχα πρόταση περικοπή. Η Γαλλία έχει εκφράσει και η γερουσία της Γαλλίας έχει εκφράσει σαφώς την ε, αντίθεσή της στα προγράμματα αυτά, στα σχέδια αυτά από την αρχή. Αν θέλουμε νέε ε, πολιτικές ε, προτεραιότητε, χρειάζεται να ιεραρχήσουμε τι δράσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά η πολιτική συνοχή και η πολιτική γεωργίας είναι παραδοσιακέ πολιτικέ όπω αναφέρθηκε επίση προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταργηθούν πλήρω οι επιστροφέ. Το τέλο λοιπόν των επιστροφών, το οποίο είναι προφανώ ένα θέμα πάρα πολύ ευαίσθητο, θα αποτελέσει προτεραιότητα για να δούμε την κλίτα κατανομή των εισφορών των εθνικών κρατών μελών. Η Φιλανδική Προεδρία είχε προτείνει τον προηγούμενο Δεκέμβριο ένα νέο κουτί, διαπραγματεύσεων, το οποίο ήταν ικανοποιητικό σε πολλά θέματα, σε ό,τι αφορά το θέμα τη άμυνα, για παράδειγμα όπου προτείνονταν ε, μείωση κατά το ίμιση. Είμαστε απόλυτα αποπισμένοι ότι αυτό που δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε και δεν θα τα δαπανίσουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να τα δαπανίσουμε σε κάθε εθνικό προπολογισμό. Και κυρίως ό,τι αφορά θέματα κρίσιμης σημασία. Ε, η έρευνα, η ανάπτυξη, η άμυνα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν αντικαθιστά αυτά που θα πρέπει να κάνουμε με λιγότερο αποτελεσματικό τρόπο σε επίπεδο κρατών μελών, σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την πολιτική για το διάστημα. Έχουμε όλοι η υπόψη μας ότι θέλουμε να πετύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά προγράμματα όπως ο Γαλιλαίος, ο Κοπέρνικος που μας δίνουν μια κάποια αυτονομία, μια κάποια ανεξαρτησία στα θέματα αυτά. Αλλά παρόλα αυτά η πρικοδότηση είναι πολύ περίπλοκη γιατί ο, το νούμερο βασίλειο ήταν βασικό εισφορέα και αποτέλεσε μεγάλη ε, απώλεια πόρων. Ύψους 10 δις υπολογίζεται. Και αυτό σε ό,τι αφορά τις εθνικές συνεισφορές θα πρέπει να την κρατήσει Μιλάμε για τη Γαλλία 7 δις ε, ευρώ αν γίνει αποδεκτή η πρόταση η της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, 9 δις αν ήταν αποδεκτή η πρόταση του 1,3% του ΑΕΠ. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε από την γερουσία της Γαλλίας να καθοριστεί ένα πιο φιλοδόξο επίπεδο δαπανών σε ό,τι αφορά και τις ε, προτεραιότητες που υπάρχουν και ε, επιδεικνύοντας ρεαλισμό. Επίσης η γαλλική γερουσία ε, λυπάται που υπάρχει τέτοια έλλειψη φιλοδοξία σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά αυτά μέσα σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα, για παράδειγμα. Ακόμα και αν ο στόχος της δημοσιονομικής σταθεροποίησης δεν είναι κάτι που μας βρίσκει σύμφωνος, θεωρούμε ότι θα πρέπει να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις του μέλλοντος και σε ό,τι αφορά και την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, η έγκριση του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου αυτού αποτελεί μια επιπρόσθετη πρόκληση. Θα πρέπει να καθορίσουμε και το επίπεδο της εμπιστοσύνης που θα έχουν σε εμάς οι πολίτες για το μέλλον. Uh, uh, ευχαριστούμε. Ο τελευταίος μας ομιλητής είναι ο κύριος Άντρε Μπένεσικ, ο ε, επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για ε, Ευρωπαϊκές Υποθέσεις ε, της, της κάτω βουλής του της Τσεχίας. Με ευχαριστώ, ε, Πρόεδρε. Λέω μιλητή. Ε, επειδή έχω προετοιμάσει την ομιλία μου στα τσεχικά, θα μιλήσω σε αυτή τη γλώσσα, αν μου το επιτρέπετε. Ευχαριστώ. Ε, συνήθως σε συνεδριάσεις όπως αυτήν έχουμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν ε, το Brexit ως το κυριότερο ζήτημα και αυτό πράγματι είναι σημαντικό γιατί για παράδειγμα 25% ε, των ε, αμυντικών μας ε, δυνατοτήτων μειώνονται με το Brexit, όπως μειώνονται και σε σημαντικό βαθμό οι αμυντικές μας τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες πλέον. Από εκεί και μετά υπάρχουν μία σειρά από προκλήσεις στο δημοσιονομικό επίπεδο που προέρχονται από το Brexit. Ωστόσο, το Brexit δημιουργεί και κάποιες ευκαιρίες, ευκαιρίες δηλαδή που μπορούν να δώσουν όθηση για τον εξυγχρονισμό της Ένωσης θα χρειαστεί δηλαδή τώρα μια αναδιάρθρωση, αν θέλετε, των οικονομικών μας. Ε, και βέβαια ε, ο εξυγχρονισμός στον οποίο αναφερόμαστε δεν θα πρέπει να αποτελέσει αυτό σκοπό. Θα πρέπει να ενσωματωθεί μέσα στο πολυμετές δημοσιονομικό πλαίσιο, έτσι ώστε αυτό με τα κατάλληλα κονδύλια να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τις μελλοντικέ μας προκλήσεις και προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελέσει ένα σημαντικό παγκόσμιο ε, παίκτη. και βλέπουμε πώς οι νέες προκλήσεις λαμβάνονται υπόψη ε, στο πολιτές του νοσονομικού ε, ε, πλαίσιο. Για παράδειγμα, το ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι δαπάνε σε ό,τι αφορά την νεολαία, για παράδειγμα, το ζήτημα του ασύλου, η αύξηση των δαπανών ταυτόχρονα και για την έρευνα και για την καινοτομία ή και τον τομέα της ασφάλειας. Έχουμε λοιπόν εδώ να κάνουμε με τομεί ε, στους οποίους η καινοτομία αποτελεί κάτι το εξαιρετικό σημαντικό και αυτό βέβαια ισχύει ιδιαίτερα ε, για, ε, για τις ανεπτυγμένες χώρες. Εμείς ως Τσεχία Ε, συγκαταλεγόμασταν στις 10 ε, πιο βιομηχανισμένες χώρες της Ευρώπης ανάμεσα στους δύο ε, παγκοσμίους πολέμους. Τώρα βρισκόμαστε σε μια φάση περαιτέρω ανοικοδόμησης βέβαια και χρειαζόμαστε βέβαια και να υποστηρίξουμε από τη μία πλευρά την σλοβακική μας οικονομία αλλά από την άλλη πλευρά να υποστηρίξουμε την κοινοτομία για τις επιχειρήσεις μας. Θα πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε τις εργασίες μας, ε, ό,τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα να ε, προσανατολίζεται ε, προς το μέλλον, χωρίς όμως να ξεχάσουμε τις παραδοσιακές μας πολιτικέ, πολιτικές, δηλαδή την αγροτική πολιτική και την πολιτική συνοχής. Καθώς οι εν λόγω αυτές οι πολιτικές δεν έχουν υπεραξία, αν θέλετε, μόνο οικονομική, αλλά και κοινωνική. Και επιχαίρουμε το γεγονός ε, ότι ακριβώς η τσεχική ε, Προεδρία του Συμβουλίου θέλει να επιτύχει αυτή την ισορροπία ανάμεσα στις πιο παραδοσιακές, αν θέλετε, ε, πολιτικές της Ένωσης, αλλά και τις πολιτικές για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων. Η κοινωνική μας ευημερία συνάδει ε, με την οικονομική μας ε, ε, ευημερία και βέβαια πρέπει να έχουμε και το απαραίτητο πλαίσιο ασφάλειας. Το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να καλύψει τα πάντα. Χρειαζόμαστε δηλαδή και διασφάλιση σε αυτό το επίπεδο και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και χρειαζόμαστε και τον κατάλληλο μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων. Έχουμε ήδη μία σειρά από αποστολές και έξι στρατιωτικέ αποστολέ ε, Έχουμε για παράδειγμα 2.000 συνολικά ε, άτομα στο προσωπικό της Ένωσης ε, και 3.000 στρατιωτικό προσωπικό που βρίσκονται αποσπασμένοι σε μία σειρά από χώρες, ενώ έχουμε αναλάβει και τον ηγετικό ρόλο στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών σε μία σειρά από αυτές τις αποστολές. 1,5 εκατομμύρια άτομα γενικά απασχολούνται στο ε, πλαίσιο ακριβώ τη ηγεσία εδώ ε, του ηγετικού ρόλου που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, το συνολικό κονδύλ εδώ ανέρχεται στα 200 δι ευρώ. Οπότε ακριβώς επειδή παίζουμε ένα τόσο σημαντικό ρόλο εδώ, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε και άλλες χώρε και άλλους φορείς οι οποίοι τάσσονται υπέρ της αύξηση τη ασφάλεια ανά τον κόσμο, όπω οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Θα πρέπει δηλαδή να έχει ε, το ΝΑΤΟ και ε, την, ε, τις κατάλληλες ικανότητες ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει και αποτρεπτικά. 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν ταπανηθεί προς αυτή την κατεύθυνση και γι' αυτό ακριβώς και εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούμε ένα πολύ σημαντικό εταίρο του ΝΑΤΟ. Βέβαια και το νέο κεφάλαιο για το περιβάλλον και για το κλίμα του πολιτού είναι πολύ σημαντικό γιατί θέλουμε να καταστούμε ως Ευρώπη η πρώτη ήπειρος που θα επιτύχει την κλιματική ουδετερότητα και για να το πετύχουμε αυτό θα χρειαστούμε τις απαραίτητες επενδύσεις ε, στην έρευνα, στην ε, καινοτομία και θα πρέπει να υποστηρίξουμε κατάλληλα και την βιομηχανική αναπροσαρμογή. Αυτές λοιπόν θα πρέπει να αποτελέσουν τις απόλυτες προτεραιότητές μας. Και για μας ως Τσεχία προφανώς είναι σημαντικό να επιτύχουμε βελτίωση της ευημερία μας, αλλά ταυτόχρονα ε, θα πρέπει να επιτύχουμε και την ε, τους ε, περιβαλλοντικούς στόχους που έχουμε θέσει. Και για να το κάνουμε αυτό, όπως είπαμε, πάντο θα πρέπει να συνοδεύεται η προσπάθειά μας από την ε, επένδυση στην καινοτομία. Και θα πρέπει αυτή η προσπάθεια να λάβει παγκόσμιο χαρακτήρα, γιατί σε διαφορετική περίπτωση ό,τι και αν κάνουμε εμείς εδώ, όλη η παραγωγή θα μετεκατασταθεί πολύ απλά στην Κίνα. Στην Κίνα δηλαδή, όπου τα πρότυπα είναι πολύ χαμηλότερα σε περιβαλλοντικό επίπεδο. Έτσι βέβαια με αυτόν τον τρόπο δεν θα βελτιωθεί τίποτα σε ό,τι αφορά το περιβάλλον παγκοσμίω. Ο κύριο ε, Ντόμαγκο μιλώσευε, τώρα έχει ε, το λόγο από την Κροατία. Παρακαλώ, δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Γνωρίζουμε ε, πολύ καλά πως η χρηματοδότηση τη Ένωση και ο προπολογισμό τη Ένωση αποτελούν σημαντικά ζητήματα για όλα τα κράτη-μέλη, είτε για τα κράτη-μέλη που λαμβάνουν περισσότερα κρατη και που δαπανούν περισσότερα. Και Ε, το να μην έχουμε τα κατάλληλα κονδύλια ουσιαστικά έχει το, το αντίθετο αντίκτυπο, δηλαδή αυξήνει τον ευρωσκεπτικισμό. Ε, Αντιθέτω, λοιπόν, ο προπολογισμό αυτό μπορεί να αποβεί προ όφελο όλων των κρατομελών εφόσον αξιοποιείται με τον κατάλληλο τρόπο, δηλαδή την ε, αξιοποίηση των κατάλληλων υπηρεσιών, αλλά και ε, το, την, το να διασφαλίζουμε ότι οι επιχειρήσει οι οποίε αποφελούνται έχουν την έδρα του στην Ένωση και ανήκουν ε, στη, στην Ευρώπη. Επίσης ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, τις δημογραφικές εξελίξεις και την ε, μαζική διαρροή των νέων μας πως τις πλουσιότερες χώρες τα πλουσιότερα κράτη-μέλη. Αν θέλουμε λοιπόν να παραμείνει συνεκτική η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας πως η μετανάστευση έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις και σε οικονομικό και σε κοινωνικό και σε πολιτικό επίπεδο. Και ε, σε πιο ταμακτικό βέβαια επίπεδο αυτές οι επιπτώσεις γίνονται αισθητέ στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Εδώ θα πρέπει να είμαστε λοιπόν ταχύτεροι στην ε, ανταπόκρισή μας ε, και πιο έξυπνοι και ταυτόχρονα θα πρέπει να έχουμε πάντοτε κατά νου την οικονομική ράχο κοκαλιά αν θέλετε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κινητήρα της οικονομικής ανάπτυξης που είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν θα πρέπει θεωρούμε να επιτηρεί το πόσο ε, μεγάλο είναι το κομμάτι των κονδυλίων ε, που κατευθύνεται προ το δημόσιο τομέα και ποιο είναι το κομμάτι που κατευθύνεται στον ιδιωτικό τομέα και ιδιαίτερα στι μικροπεσαίε επιχειρήσει προκειμένου να δαπανούμε με σοφία αυτά τα κονδυλία. Θα πρέπει δηλαδή να διασφαλίσουμε ότι μέσα στι ε, επόμενε δεκαετίε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πιο σύγχρονη, πιο φιλοπιλωτική, πιο ανταγωνιστική και σε παγκόσμιο επίπεδο πιο ολοκληρωμένη αν θέλετε. Η κυρία Βαμποσά τώρα από το Βέλγιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και θα μιλήσω Ολλανδικά. Και θα ήθελα να πω καταρχάς ότι είμαι χαρούμενη που σας βλέπω και από μια άλλη πλευρά και είμαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πέρα από την ε, Βελγική Βουλή. Θα ήθελα να τονίσω μερικά στοιχεία. Καταρχά, είναι για μα πολύ σημαντικό το γεγονό ότι δεν θα υπάρξει αύξηση των ε, εθνικών εσφορών γιατί με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου έχει περιοριστεί ο προπολογισμό ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να προσαρμοστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά τα τελωνιακά έσοδα, άκουσα και τη συζήτηση που έγινε για τους ιδίους πόρους και τους καινούργιους ιδίους πόρους. Για μια εμπορική περιοχή όπως η Φλάνδρα, αυτά τα τελωνιακά έσοδα είναι πολύ σημαντικά και δεν συμφωνούμε αυτό που αναφέρεται για το ποσοστό το οποίο θα πρέπει να άμα κρατούν τα κρατημέρια θα πρέπει να μειωθεί από το 20% στο 10% στο ίμιση και κάτι άλλο τελευταίο και σημαντικό στοιχείο το, Ευρωπαϊ... το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στη σημερινή κατάσταση θα πρέπει να επωφεληθεί για να μεταρρυθμίσει διάφορα θεσμικά όργανα σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τον μηχανισμό κατανομής, αυτό το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Αυτό δεν λαμβάνει υπόψη ε, τον αντίκτυπο του Brexit σε διάφορες ευρωπαϊκές περιοχές. Θα πρέπει να φροντίσουμε το ταμείο αυτό να αναθεωρηθεί, να προσαρμοστεί, προκειμένου να υπάρχει προσαρμογή και στις μελλοντικές καταστάσεις, γιατί το θέμα είναι να υπάρχει πιο δίκαιη κατανομή των μέσων. Και τέλος ε, δεν ε, συμφωνούμε με το γεγονό ότι σήμερα 40% του ευρωπαϊκού προπολογισμού πάει στη γεωργία. Ναι, έχουν προβλήματα οι γεωργοί και θα πρέπει να βοηθηθούν, αλλά Τελικά τα χρήματα αυτά σε πολλέ περιπτώσει καταλήγουν σε μεγάλε βιομηχανικέ ε, γεωργικέ εκμεταλλεύσει που δεν χρειάζονται τέτοιου είδου ενισχύσει. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει ένα άνωτατο όριο και να δαπανίσουμε τα χρήματα αυτά σε καλύτερου ε, σε καλύτερε μέρη, όπω για παράδειγμα η έρευνα και η ανάπτυξη. Ευχαριστώ πολύ. Από την Πορτογαλία, ο Παύλο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θεωρώ πως ε, είναι πολύ σημαντικό πρωτό ορίσουμε τον προπολογισμό και το πώς θα καταναμηθεί, ε, να ορίσουμε τις προτεραιότητές μας, τις στρατηγικές μας. Ε. Και προφανώς λοιπόν δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε να έχουμε μια καταγερματισμένη Ευρώπη. Δηλαδή θα πρέπει η εξόχως σε περιοχές ε, είδαμε ε, πως υπήρξε μια ε, προσπάθεια να αποκλειστούν από το Ταμείο της Δίκαιος Μετάβασης. Το, κάτι τέτοιο δεν είναι σωστό. Από εκεί και μετά η αύξηση του ποσοστού της χρηματοδότησης που ζητήθηκε θεωρούμε πως ουσιαστικά υπονομεύει την, την, την κατάσταση αυτών των ε, περιοχών που ήδη αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα στο να επιτύχουν την κατάλληλη ε, επίπεδο ε, συνοχής με τις υπόλοιπες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. δεν θα ήθελα να ε, ξεχάσω το, ε, να, να, να, να παραμιλήσω το γεγονός ότι θα πρέπει να ε, έχουμε τις απαραίτητες επενδύσεις στο τομέα της, της έρευνας και της τεχνολογίας, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να επιτύχουν την μετάβαση ειδικότερα και στο ψηφιακό επίπεδο. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω βλέπω ότι ορισμένες από αυτές τις ε, στρατηγικές ουσιαστικά μεώνονται προς όφελος ε, κάποιων ε, άλλων πολιτικών, πράγμα όμως που δεν θα πρέπει να λάβει χώρα, δηλαδή πολιτικές όπως η αγροτική πολιτική, πολιτική αλλιάς και ούτω καθεξής. Όχι, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βρει νέες επίγες χρηματοδότησης και όχι να θέσει σε κίνδυνο τις ήδη υφιστάμενες εντρεωμένες πολιτικές. Δεν μπορεί λοιπόν να απολέσει το κεντρικό και ηγετικό ρόλο που παίζει ε, τη σήμερα η Ένωση στον κόσμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο ε, Λεβαντόφσκι. Ένα πρώτο ζήτημα που θα ήθελα να θέσω είναι ότι δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον ε, προπολογισμό της Ένωσης ως την πανάκια που θα λύσει όλα τα προβλήματα της Ένωσης. Μόνο το 2,5% από της Ένωσης καλύπτει. Όμως έχει εδώ μπορεί να ασκήσει πραγματικά σημαντικό ρόλο. Ένα δεύτερο στοιχείο που θα ήθελα να αναφέρω είναι ε, το πώς μπορούμε, είπαμε εδώ, να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες προκλήσεις ε, μέσω του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου. Τα όσα είπαμε σήμερα εδώ δεν έχουν να κάνουν ούτε με τις παγκόσμιες προκλήσεις, ούτε με τον ηγετικό ρόλο της Ευρώπης. Άρα, οι πολιτικοί μας ηθήνοντε θα πρέπει και καλούνται να λάβουν ρεαλιστικέ ε, αποφάσεις και όλοι αναμένουν ε, να, ε, ε, να, να λάβουν κάποια δώρα, αν θέλετε, τη τελευταία στιγμή από τον κύριο Μισελ. Το Ευρωπαϊκό λοιπόν Κοινοβούλιο βρίσκεται σε μια δυσάρεστη θέση αυτή τη στιγμή, όπου απλά βρίσκεται σε στάση αναμονής από το Μάιο του 2019 παρακολουθώντα τον κύριο Μισελ, ουσιαστικά να ευθυγραμμίζεται περισσότερο με τη στάση των κρατών μελών εκείνων που συνεισφέρουν περισσότερο στον προπολογισμό των έντων. Ήδη λοιπόν ε, έγινε μια προσπάθεια και μάλλον θα, ακολουθήσει, θα ακολουθήσουν και άλλε προσπάθειε να ασκηθούν πολύ σημαντικέ πιέσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ουσιαστικά δηλαδή ε, αυτό συνέβη και την τελευταία φορά. Δηλαδή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου μας ασκείται ε, πολύ μεγάλη πίεση ακριβώς ε, χρόνου και ουσιαστικά η μοναδική φορά που μπορέσαμε να έχουμε αύξηση των κοντιλίων του προεδρικού του δημοσιονομικού πλαισίου ήταν την περίοδο 2005 με 2013 που επιτύχαμε αύξηση μόνο κατά 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε ε, αυτή την περίοδο σε μια πολύ δύσκολη θέση εκτός και αν συμβεί κάποιο θαύμα. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος, ο κύριος Μάσιμο Καραβάνια από την Ιταλία. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Έχουμε πολύ, τρεις πολύ απλές ερωτήσεις. Ε, το πρώτο που κάνει κανείς όταν του λείπουν πόροι είναι να μειώσει το κόστος ε, και θα πρέπει να δείτε ουσιαστικά ε, τι αποκομίζεται από το spending review, από την επισκόπηση των δαπανών. Όταν υπάρχει κρίση, είναι αδύνατο να πάει κανείς να ζητήσει από τα κράτη που συνεισφέρουν καθαρά να αυξήσουν τη συνεισφορά τους. Αυτό δεν είναι δυνατόν να συμβεί. Τη στιγμή της κρίσης είναι αυτονόητο. Το τρίτο θέμα σε ό,τι αφορά την ε, φορολογική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Μιλάμε για ε, το φόρο επί των πλαστικών. Θέλουμε να καταλάβουμε καλύτερα σε τι συνιστατέ, γιατί αν κατάλαβα καλά αφορά μόνο τα πλαστικά που δεν έχουν ανακυκλωθεί και θα πρέπει να μπούμε σε λεπτομέρειες. Στην Ιταλία έχουμε ένα παράδειγμα ενός τέτοιου φόρου επί πλαστικών και είχε πολύ αρνητικό αντίκτυπο. Ε, δηλαδή, ε, επευλήθη αυτός ο, ο φόρος στις πρώτες ύλες, ε, στην παραγωγή και είχαμε κατάρρευση του τομέα το Δεκέμβριο κατά 7,2%. Θα είναι αρνητικό ο αντίκτυπος. Ε, δηλαδή, είναι μεγαλύτερο το εισόδημα που χάνεται κατά τη ε, διάρκεια της παραγωγής ε, παρά τα όσα αποκομίζονται από το φόρο. Δηλαδή είναι εντελώ ανόητος ο φόρος αυτός. Τελευταία ερώτηση, απλούστευση. Δεν σκεφτήκατε ποτέ να πλουστεύσετε τον προϋπολογισμό. Τελικά αν έχουμε καθαρούς συνεισφέροντες, δεν μπορούν ε, μόνο να συνεισφέρουν αυτοί και κατόπιν να έχουμε τις πολιτικές που αποφασίζει το Κοινοβούλιο με τους ίδιους πόρους. Oh. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Άνταμ Κάλους από την Τσεχική Δημοκρατία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω τη μητρική μου. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να υποστηρίξω τη θέση της κυβέρνησης της Τσεχίας, να τονίσω ότι ο μελλοντικό προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι ισορροπημένο. Θα πρέπει να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ παραδοσιακών και νέων πολιτικών. Αν μιλάμε για πιθανές περικοπές, δεν θέλουμε περικοπές σε παραδοσιακές πολιτικές. Να σας υπενθυμίσω ότι η τσεχική δημοκρατία έδωσε ιδιαίτερα έμφαση στην πολιτική συνοχής και στην κοινή αγροτική πολιτική. Θέλουμε επίσης να έχουμε καλές προϋποθέσεις για την εφαρμογή των πολιτικών αυτών. Όλες οι χώρες στην ομάδα των φίλων της συνοχής υποστηρίζουν την ιδέα να διατηρηθεί η πολιτική συνοχή όσο έχει αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι μπορούμε να δούμε ότι η πολιτική συνοχή μας βοηθά να βελτιώσουμε τη σύγκληση μεταξύ των χωρών. Είναι και σημαντική για την εσωτερική αγορά. Πρέπει να διατηρήσουμε το επίπεδο επενδύσεων. Επομένω, η Τσεχία δεν μπορεί να δεχτεί μείωση των επιδοτήσεων. Η πολιτική συνοχής θα είναι αποτελεσματική μόνο αν τα κράτη-μέλη έχουν περισσότερε αρμοδιότητε όταν θα αποφασίζουν ε, για το ποιε είναι οι επενδυτικέ του προτεραιότητε. Παραδείγματο χάρη, τα κράτη-μέλη θα ήθελαν να έχουν μεγαλύτερη ελευθερία για να μεταφέρουν πόρους ε, μεταξύ των διάφορων ταμείων. Και τώρα, σε ό,τι αφορά την αγροτική πολιτική, υποστηρίζουμε μόνο εκούσια ανώτατα όρια των άμεσων πληρωμών. Οι αλλαγέ θα πρέπει να γίνουν μόνο σε χώρε που ξεπερνούν τα όρια. Σε ό,τι αφορά τώρα τα έσοδα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι το σύστημα ιδίων πόρων θα πρέπει να είναι δίκαιο, διαφανέ και αποτελεσματικό και δεν θα πρέπει να προκαλεί προβλήματα στα λιγότερο αναπτυγμένα κράτη-μέλη φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία στο σύστημα των ιδιοπόρων. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να διατηρήσουμε το σημερινό σύστημα και να, να προσπαθήσουμε να το απλουστεύσουμε. Να ζητήσω επίση από την κροτική Προεδρία να δράσει ως ένας έντιμος διαμεσολαβητής και να βρει μια συμβαστική λύση. Ξεπεράσατε υπερβολικά το χρόνο, λέει ο πρόεδρο. Κυρία Σαμπίν Τίλε, από τη Γαλλία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως ε, καταλάβατε και είπαν κάποιοι συνάδελφοι, για τη Γαλλία η έννοια της ευρωπαϊκής κυριαρχίας είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και αν δούμε τον προπολογισμό που μας προτείνεται, βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές περικοπές στον προπολογισμό σε θέματα που συνεισφέρουν στην κυριαρχία μας και είναι παράδεκτα παράδειγμα στις αν δούμε την νέα αγορά, την καινοτομία και τα ψηφιακά, παρά ε, το ότι οι ηγέτε των κρατών τοποθετήθηκαν ε, υπέρ των μελλοντικών τεχνολογιών και υπέρ των επενδύσεων, ε, συνεχίζουν να χρησιμοποιούν αυτά τα κονδύλια ως περιθώριο λιγμών. Επίσης, αν δούμε τι συμβαίνει στην ΚΑΠ και στη μείωση των ευρωπαϊκών κονδυλίων στον τομέα της άμυνας, όλα αυτά είναι θέματα τα οποία αποτελούν προτεραιότητα για να εγκαθιδρύσουμε την ευρωπαϊκή κυριαρχία. Ε, ε, βλέπουμε να υπάρχουν δύο φιλοσοφίες σήμερα. Υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη που δεν θέλουν να αυξηθεί ο προπολογισμό, ε, να θέλουν να είναι σταθερός ο προπολογισμό και θέλουν να δράσουν έτσι ώστε οι προτεραιότητες να εντάσσονται στον προπολογισμό και θέλουν άλλοι να έχουν ως αφετηρία τις προτεραιότητες και να δουν πώς θα τις χρηματοδοτήσουν. Είναι λοιπόν μια σημαντική απόφαση αυτή που θα πρέπει να ληφθεί και θα πρέπει να δούμε και τη μέθοδο. Πώς ε, θα κατορθώσουμε να τα χρηματοδοτήσουμε όλα αυτά, αλλά φυσικά <laughs> συνάδοντας και με τον προπολογισμό, σε σχέση με τον προπολογισμό των κρατών μελών. Ε, δεν νομίζω ότι πρέπει να αποσυνδέσουμε τον ευρωπαϊκό προπολογισμό από τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Ε, νομίζω ότι στο επίπεδο αυτό θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη, μεγαλύτερος συσχετισμός. Ευχαριστώ κυρία Άννα Μπονφρίσκο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολλές φορές είχα την ευκαιρία να πάρω το λόγο στις εργασίες της Επιτροπής μας σε σχέση με τις ε, ισχυρές ανησυχίες που θα πρέπει να έχει η Ευρώπη σε σχέση με την γεωπολιτική θέση που θα λάβει και φυσικά αυτό έχει να κάνει και με τις ε, κύριες ε, οικονομικές δραστηριότητες αλλά και με τον προπολογισμό της. Γι' αυτό εμείς θεωρούμε πολύ επικίνδυνη οποιαδήποτε περικοπή τη χρηματοδότησης ε, στην κοινή αγροτική πολιτική γιατί θεωρούμε ότι πολύ σύντομα θα μπορούσε να γίνει ένα από τα στοιχεία που θα είναι ε, κατεπήγοντα στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμία. Αλλά προσπαθώντα να βρούμε ένα σημείο ισορροπία για του νέου πόρου και για του ίδιου πόρου που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να υιοθετήσει μέσω νέας φορολόγησης. Εμείς ε, είμαστε αντίθετοι σε όλα αυτά. Αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο σήμερα είναι να αναπτύξουμε κάποιες σκέψεις, κάποιους προβληματισμούς, όπως αυτές που ακούστηκαν από κάποιους συναδέλφους από το Τσεχικό Κοινοβούλιο, παραδείγματος χάρη, για τη συνοχή ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δυστυχώς σε πάρα πολλά ε, σημεία έχει αποτύχει και αυτό το λέω εκπροσωπώντας ε, μία χώρα ιδρυτή. Πολύ λίγο αποτελεσματική ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα αυτό. Εγώ δεν είμαι πεπισμένη ότι υπάρχει προσθεμένη αξία για τις χώρες από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει φτάσει στο ωριά της σήμερα και πολύ γρήγορα θα πρέπει να βρει νέους ε, ε, τρόπους ε, οικονομικού προγραμματισμού και νομίζω ότι το κύριο πρόβλημα είναι το θέμα της άμυνας και της ασφάλειας. Και η ερώτησή μου είναι η εξή. Τι σκέφτεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει χωρίς να χάσει περαιτέρω χρόνο σε σχέση με τις δαπάνες για την αμυντική βιομηχανία που αυτή ε, ουσιαστικά κυριαρχούσε ε, στις ε, εποχές της οικονομικής άνθησης και για την προστασία των Ευρωπαίων πολιτών, για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών. Ο κύριος Φερνάντο Αναστάζιο από την Πορτογαλία. Θα μιλήσω στα πορτογαλικά. οι διαπραγματεύσει για το πολιτιστικό δημοσιονομικό πλαίσιο ε, θα είναι δύσκολε, ε, Δηλαδή 27 κράτη-μέλη προσπαθούν να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα ε, το οποίο προήγηψε με το Brexit, δηλαδή μείωση του προπολογισμού κατά 60 κατά όλη αυτή την περίοδο και βέβαια ε, εδώ το ζητούμενο είναι να βρεθούν νέε λύσει προκειμένου να επιτύχουμε την υλοποίηση τη αντίστοιχα για την βιώσιμη ανάπτυξη. Και βέβαια προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τι διάφορε πολύπλοκε προκλήσει που αντιμετωπίζουμε ω Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω να φτάσουμε σε μια συμφωνία ε, ε, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα είχαμε πρόβλημα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουμε και σε πρακτικό επίπεδο και σε πολιτικό επίπεδο και προκειμένου να αντιμετωπίσουμε νέε προκλήσει. Θα πρέπει λοιπόν να προσεγγίσουμε αυτέ τι διαπραγματεύσει με αισιοδοξία, ε, προκειμένου να φτάσουμε σε μια συμφωνία με αποφασιστικότητα και σε ένα αποτέλεσμα το οποίο ε, θα γίνει αποδεκτό από όλου. Ε, τώρα, κατά την άποψη τη σοσιαλιστική ομάδα από την πλευρά τη Πορτογαλία, θέλουμε αυτή η συμφωνία να επικεντρωθεί σε ορισμένα βασικά ζητήματα τα οποία θα αναφέρω σύντομα. Θα πρέπει το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο δηλαδή να παραμένει γύρω στο 1,16% του δηλαδή στο ε, επίπεδο της δέσμευσης που ανέλαβαν όλα τα κράτη-μέλη. Και επίσης το νέο πρωτεύουσα πλαίσιο να, να, να ανταποκρίνεται στις ε, φιλοδοξίε τη Ευρώπη σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση τη κλιματική αλλαγή, ε, την ε, ψηφιακή μετάβαση, ε, το ζήτημα τη ασφάλεια και άλλα. Και βέβαια, οι πολιτικέ όπω η κοινή αγροτική πολιτική δεν θα πρέπει να αποτελέσουν μεταβλητέ εδώ. Θα πρέπει δηλαδή η ανταγωνιστικότητα, η συνοχή και η ανάπτυξη να παραμείνουν ω βασική άξονα. Και θα πρέπει να συνεχίσουμε την διαδικασία εμπάθηση τη ενοποίηση τη Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση τη Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαι πεπισμένο ότι θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε με επιτυχία ε, αυτό το εγχείρημα. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριο Αντρέ Μέρεγια από τη Γερμανία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Επανέρχομαι σε μια περιγραφή που κάνατε στην αρχή της ομιλίας σας. Είπατε ότι δεν μπορούμε δηλαδή ε, σε ό,τι αφορά αυτέ τι διαπραγματεύσει, ουσιαστικά να εγκαταλείψουμε κάποια βασική προτεραιότητα που είχαμε και να υιοθετήσουμε μία άλλη. Εκείνο που θα έλεγα εγώ ε, ήταν, θα ήταν ε, να αξιοποιήσουμε κατά κάποιο τρόπο τι ε, προτεραιότητε για να βοηθήσουμε περισσότερου ανθρώπου. Δηλαδή κατά δική μου άποψη το ζήτημα δεν είναι απλώ και μόνο να έχουμε περισσότερα κονδύλια αλλά να υπάρχει πολιτική βούληση και την κατάλληλη εφαρμογή των σχετικών προτεραιοτήτων. Ε, και να πω βέβαια ότι αυτό το πολιτιστικό δημοσιονομικό πλαίσιο ε, αναφέρεται σε 280 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή σε κάτι το πολύ μεγαλύτερο από ότι ένα μεμονωμένο ε, προπολογισμό σε κράτου μέλου. Άρα λοιπόν θα πρέπει ε, και το ζήτημα του Brexit, για παράδειγμα, να το αντιμετωπίσουμε και με περισσότερα κονδύλια και ανακατανομή των σχετικών κονδυλίων. Υπάρχουν ε, ε, κάποιοι τομεί ε, σε σχέση με του οποίου ζητήθηκαν περισσότερα κονδύλια. Το Green Deal, για παράδειγμα. Τέθηκαν πολλά ερωτήματα. Ένα δισεκατομμύριο για όλα αυτά τα χρόνια με το ίμιση να αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το υπόλοιπο να έχει κατανεμηθεί. Τι σημαίνει αυτό, 15 δισεκατομμύρια δηλαδή ευρώ ετησίω των προπολογισμών. Από πού πρέπει προέρχονται αυτές οι, αυτή η χρηματοδότηση. Δηλαδή εμείς όταν έχουμε ακόμα και αύξηση της ε, δικής μας συνεισφοράς κατά 0,1% και μόνο μιλάμε για 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Οπότε ε, ε, τίθεται το ερώτημα από πού θα προέλθουν αυτά τα κονδύλια γιατί τελικά έρχονται από τα κράτη-μέλη. Και βέβαια επανέρχομαι σε αυτό που αναφέρθηκε, ότι δηλαδή θα πρέπει να επιτύχουμε την αποδοχή της Ένωσης από τους πολίτες, αλλά αυτό δεν θα το επιτύχουμε με το να δημιουργήσουμε έλλειμμα στα δημόσια οικονομικά των κρατών μελών. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα ε, στα ζητήματα εκείνα τα οποία τελικά αντιμετωπίζονται με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο σε επίπεδο, ε, στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και υπάρχουν πολλά παραδείγματα ε, για τέτοιου είδου παρεμβάσει. Ε, θεωρώ πως θα πρέπει να φτάσουμε στο επίπεδο της ε, χρηματοδότησης του στάξης του 1% ε, του εθνικού εισοδήματος. Από εκεί και μετά σε ό,τι αφορά το σύστημα των ιδίων επών, θεωρώ πως θα πρέπει να το εξετάσουμε περαιτέρω, ειδικότερα δηλαδή σε ό,τι αφορά αυτό το επιχείρημα για την αρχή του κράτους δικαίου και για την συγκέντρωση αυτών των πόρων. Εντάξει, αυτά είναι κάποιες από τις βασικές σκέψεις που έχω κάνει δεν έχω παραπάνω χρόνο στη διάθεσή μου, απλώ θα ήθελα να επαναλάβω αυτό που είπα στην αρχή, ότι δηλαδή θα πρέπει οι νέε μα προτεραιότητε να μην υποκαταστήσουν παλαιότερε. Ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ. Θα μιλήσω ισπανικά. Ο προεπιλογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αφήσει πίσω ούτε άτομα ούτε περιφέρειε, δεν μπορεί να διευρύνει τι διαφορέ μεταξύ των περιφερειών, ούτε θα πρέπει να χρησιμοποιείται Γι' αυτό το λόγο έχουμε ξεκάθαρο παράδειγμα στην Ισπανία και βλέπουμε τι σημαίνει στην Εξτρεμαδούρα, στην περιοχή μου όπου ε, οι αγρότες διαμαρτύρονται και ζητούν ε, δίκαιες τιμές ε, και μια κοινή αγροτική πολιτική να τους βοηθήσει να διατηρήσουν τις εκμεταλλεύσεις τους. Ζητούν κάτι δίκαιο, ζητούν δικαίωμα στο μέλλον και εμείς θα πρέπει να τους βοηθήσουμε να διατηρήσουν τον ήρό τους. Είναι θέμα βούλησης. πρέπει να προτείνουμε έναν οδικό χάρτη χάρτη και να θέσουμε κάποια αριθμητικά στοιχεία. Α μην επιτρέψουμε να μείνει κανεί πίσω, α μην επιτρέψουμε άντρε και γυναίκες που δουλεύουν νυχθημερών να πρέπει να σταματήσουν τι δραστηριότητέ του. Α μην επιτρέψουμε να διάσουν τα μικρά χωριά και να χαθούν ευκαιρίε. Ο προπολογισμό είναι το πιο σημαντικό εργαλείο πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι θέμα επιλογή. Ε, να επιλέξουμε, να θέσουμε προτεραιότητα σε κάποιε πολιτικέ έναντι άλλων. Μία από τι μεγάλε προκλήσει είναι ε, να δημιουργήσουμε μία σταθερή ανάπτυξη. Θέλουμε μία Ευρώπη που να αναπτύσσεται και α ε, επενδύσουμε στην ανάπτυξη, στην κοινοτομία, στην τεχνολογία αλλά ας στοιχηματίσουμε στους ανθρώπους τα προβλήματά τους, ας μην ε, τους χάνουμε από την εικόνα. Ε, ε, είχαμε ε, μεγάλο ποσοστό συμμετοχή στις ευρωεκλογέ. Μας ε, είπαν οι άνθρωποι ότι τους ε, ενδιαφέρει η Ευρώπη να ακούσει τα προβλήματά τους και α επιστρέψουμε στους πολίτες αυτές τις προσδοκίες με έναν προϋπολογισμό που να αρμόζει. Περιμένουν πάρα πολλά οι άνθρωποι από αυτόν τον προϋπολογισμό. Οι Γεωργοί, ας μην τους απογοητεύσουμε. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Μπογκδάν Τζόντσα. Ευχαριστώ και θα χρησιμοποιήσω την πολωνική γλώσσα. Για μένα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένα ορθολογικό έργο. Και μόνο ως, τότε, ως τέτοιο μπορούμε να την υποστηρίξουμε ως ομάδα ICR. Και παρατηρώ λοιπόν κάποια περίεργα φαινόμενα σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το ευρωπαϊκό λοιπόν project, κυρίε και κύριοι, θα πρέπει να το αναλύουμε διαρκώ και σε ό,τι αφορά τα αριθμητικά στοιχεία. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι σημαντικό να λέμε την αλήθεια σε ό,τι αφορά του καθαρού εισφορεί και του καθαρού ε, ε, ε, αποδέκτε τη βοήθεια. Αν Κάποιες αναλύσεις και έρευνες υποδεικνύουν ότι μια χώρα η οποία διατείνεται ότι είναι καθαρός εισφορέας ε, τελικά λαμβάνει 20 δις. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε αυτούς τους μύθους. Θα πρέπει να λάμψει η αλήθεια. Και κάτι άλλο. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε πολλά προβλήματα, Προφανώς χρειαζόμαστε και πολλούς πόρους. Αν θέτουμε νέους στόχους, αν ε, αντιμετωπίζουμε νέες προκλήσεις, θα πρέπει να ανταποκριθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Σύμφωνο με όλα αυτά που λέμε για το πράσινο σύμφωνο, για την προστασία του περιβάλλοντος και του καθεξής. Ναι, αλλά αυτά τι συνεπάγονται. Εγώ προσωπικά τα προσυπογράφω όλα αυτά. Αλλά παράλληλα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνουν χώρα και άλλε εξέλιξει, τι οποίε θα πρέπει να αναλύσουμε. Για παράδειγμα, παρακολουθώ τι συζητήσει για το πακέτο κινητικότητα και αυτό νομίζω καταδεικνύει το εξή, ότι αν τεθεί σε εφαρμογή το πακέτο κινητικότητε, εκατοντάδε χιλιάδε ε, οχήματα θα γυρνάνε άδεια στις πατρίδες τους και μιλάμε για τρία δις ε, τόνους ε, διοξιδίου του άνθρακα που θα εκλείονται από τα οχήματα αυτά. Αυτές οι εταιρείε λοιπόν θα αποτανθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποζημωθούν. Αυτά λοιπόν είναι πολύ περίεργα. Ευχαριστώ πολύ από την Κύπρο. Chairman, I will speak in Greek. Ξεκινώ την παρέμβασή μου ευελπιστώντα ότι η προσεχή ειδική σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στι Βρυξέλλε σε λίγε μέρε θα καταλήξει σε συμφωνία για το επόμενο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση των υφιστάμενων προγραμμάτων και πολιτικών τη Ένωση και η έναρξη νέων. Το νέο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να περιλαμβάνει επαρκεί πόρου για την υλοποίηση των φιλόδοξων στόχων τη Ένωση για οικολογικό και ψηφιακό μετασχηματισμό. Επίση, θα πρέπει να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τι σύγχρονε ευρωπαϊκέ προκλήσει, μεταξύ άλλων τη ραγδαία δημογραφική αλλαγή και την κύραση του πληθυσμού, τη βελτίωση των συνθηκών εργασία και τη διασφάλιση βιώσιμων συστημάτων κοινωνική προστασία και συνταξιδοτικών συστημάτων, τη δημιουργία νέων ποιοτικών και αξιοπρεπών θέσεων εργασία, την υιοθέτηση ολιστικής προσέγγιση στην αντιμετώπιση των μεταναστευτικών και προσφυγικών πιέσεων μέσω της επίδειξης έμπραχτης αλληλεγγύης και ισότιμης κατανομής βαρών μεταξύ των Ευρωπαίων εταίρων και την πρόληψη της τρομοκρατίας και εσωτερικών και εξωτερικών απειλών ασφαλείας. Περαιτέρω, θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη στόχευση των δαπανών και βελτίωση της διασύνδεσής τους με την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων με ιδιαίτερη έμφαση την υλοποίηση των στόχων βιώσιμη ανάπτυξη των ΗΕ και τη Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή. Ταυτόχρονα θα πρέπει να συμβάλλει στη βελτίωση τη ποιότητα ζωή και τη ευημερία των Ευρωπαίων πολιτών, στη μείωση του δημοκρατικού ελλείμματο και στην αποκατάσταση τη αξιοπιστία των ευρωπαϊκών θεσμών. Καταλήγοντα, θα ήθελα να τονίσω ότι η κοινή αγροτική πολιτική και η πολιτική συνοχή παρέχουν διαχρονικά πρόσθετη αξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να παραμείνουν ψηλά στι προτεραιότητε του νέου πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου μέσω τη διατήρηση του επίπεδου χρηματοδότησή του, ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά οι περιφερειακέ ανισότητε και να ενισχύεται η κοινωνική και οικονομική συνοχή. Τέλο, οι ιδιαιτερότητε των κρατών μελών τη Ένωση θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, σοβαρά υπόψη στου μελλοντικού σχεδιασμού τόσο τη κοινή αγροτική πολιτική όσο και τη πολιτική συνοχή. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Αλβάρο Αλμέδα από την Πορτογαλία. Ακούσαμε πολλές παρεμβάσεις ότι πρέπει να διατηρήσουμε την πολιτική συνεχής ε, και τις παραδοσιακές πολιτικές και την ΚΑΠ, ενώ θα χρηματοδοτήσουμε και νέες πολιτικές που αυτό θα σημαίνει ότι θα έχουμε και έναν μεγαλύτερο περιπολογισμό. Υποστηρίζω τι απόψει αυτέ και πίσω, επίσης συμφωνώ με τι ανησυχίε κάποιων ότι αυτό θα μπορούσε να σημαίνει υψηλότερους φόρους για τους Ευρωπαίους πολίτες. Αυτό δεν το θέλουμε, γιατί το να πούμε στους Ευρωπαίους πολίτες ότι πρέπει να πληρώσουν περισσότερους φόρους για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν ένας τρόπος ε, αυτοί να απορρίψουν το ευρωπαϊκό project. Εγώ θεωρώ ότι δεν χρειάζονται προσθετηφόροι για να έχουμε υψηλότερο υπολογισμό. Αυτέ οι νέε πολιτικέ σχεδιάστηκαν για να αντιμετωπιστούν παγκόσμιε προκλήσει που όλοι πρέπει να αντιμετωπίσουμε και δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Οι επιλογέ το αν θα τι αντιμετωπίσουμε σε εθνικό επίπεδο ή αν θα τι αντιμετωπίσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ε, αυτή είναι, έγκυται. Η επιλογή έγκυται για το αν θα έχουμε 27 πράσινες συμφωνίες ή μια ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία, θα έχουμε μία μεταναστευτική πολιτική, 27. Και ξέρετε γιατί οι ευρωπαϊκές πολιτικές είναι πολύ πιο αποτελεσματικές από τις εθνικές πολιτικές. Και όταν αυξάνουμε τον προπολογισμό για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις, δεν αυξάνουμε τις συνολικές δαπάνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, απλώς μεταφέρουμε δαπάνες που θα πρέπει να γίνουν σε εθνικό επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επομένως, δεν δημιουργούμε τρύπα στους εθνικούς προπολογισμού. Μειώνουμε τις εθνικές δαπάνες και έτσι δεν χρειάζεται να αυξήσετε τους φόρους για να χρηματοδοτήσετε αυτές τις δράσεις. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές χρειάζονται φρέσκο χρήμα και αυτό δεν σημαίνει υψηλότερους φόρους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Γερμανία, Κριστιαν Πετρί. sorry. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η κυβέρνηση συνασπισμού συμφώνησε ε, ότι είμαστε διατεθειμένοι ως ε, Γερμανία να αυξήσουμε την συνεισφορά στον προπολογισμό της Ένωσης. Άρα λοιπόν 13-15 ε, δισεκατομμύρια ε, θα είναι το κονδύλι το οποίο θα αυξηθεί η συνεισφορά μας λόγω του Brexit ε, και άλλων, αλλά ε, βέβαια αυτό αυτή η αύξηση δεν υπάρχει. Βέβαια θα υπάρξουν οι πολιτικοί στην χώρα μας που θα πούν όχι δεν μπορούμε να συνεισφέρουμε κάτι παραπάνω ενώ υπάρχουν πολιτικοί εδώ από την Ευρώπη που θα πούν ότι θέλουμε να επιτύχουμε την άσκηση της κοινή αγροτικής πολιτικής, της εκπαιδευτικής πολιτικής, της ασφαλείας, μετανάστευσης και ούτω καθεξής. Ε, πώς μπορούμε να το δικαιολογήσουμε αυτό όλε αυτέ τις νέε πολιτικέ ε, με λιγότερα κονδύλια. Δηλαδή προφανώ τίθεται το ζήτημα του να υπάρξουν καλύτερε συνέργειε και να υπάρξει ε, και λιγότερο φόρτο για τα την με τα όσα επιτυχάνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά από εκεί και μετά εκείνο που θέλω εγώ να πω είναι ότι δεν θα πρέπει να χάνουμε από τα μάτια μας τη συνολική εικόνα. Δηλαδή το να θέλουμε να επιτύχουμε μια νέα προτεραιότητα παρεμβολώντα την κοινή αγροτική πολιτική είναι κάτι το ασφαλμένο. Η πρόταση που έχει γίνει μέχρι τώρα από τον κύριο Μισελ αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τα μπροστά, αλλά νομίζω πως δεν θα ε, αποτελέσει αυτό, αυτή η πρόταση την τελική μας συμφωνία. Θα πρέπει δηλαδή να εξασφαλίσουμε την απαραίτητη χρηματοδότηση και ε, με εκπλήσει το γεγονό ότι ε, συζητείται τόσο εκτεταμένο το ζήτημα των ιδίων πόρων, αλλά τελικά δεν έχουμε καταλήξει πουθενά. Δηλαδή, τι θα συμβεί στην, ε, σε αυτή την περίπτωση. Απλώ σε μόνο μία συζήτηση λέμε ότι πολύ ωραίε όλε αυτέ οι ιδέε, αλλά ε, δεν θα μπορέσουμε να τι υλοποιήσουμε στην πράξη στο πλαίσιο αυτού του πλαισίου ε, και γι' αυτό ε, τα μεταφέρουμε όλα αυτά για το επόμενο ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, ουσιαστικά ε, έχει ε, εξασφαλίσει με την νομισματική της πολιτική της σταθερότητα αλλά μπορεί νομίζω πως να συνεισφέρει από τη δική της πλευρά σε μια καλύτερη χρηματοδότηση του προπολογισμού και αυτό δεν έχει ληφθεί καθόλου υπόψη στη συζήτηση μέχρι τώρα και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αντρέ Κωστόβνακ έχει τώρα τον λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, θα μιλήσω πολωνικά. Μιλάμε σήμερα για τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το έτος 2021-2027. Και μιλάμε διαρκώς ε, για δύο συγκεκριμένα στοιχεία. Δύο βασικά στοιχεία. Καταρχάς, να καλύψουμε τα κενά με το Brexit. Και κατά δεύτερον, να μιλάμε διαρκώς για περιορισμό των δαπανών σε ό,τι αφορά κάποιες ε, πολιτικές του προπολογισμού. Αυτή η συζήτηση όμως ε, βασίζεται και στην επιθυμία να σκεφτούμε από πού προέρχονται τα μέσα τα οποία δαπάνονται στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ προτού ορίσουμε τα όρια σε κάποιους πολιτικούς τομείς και πολύ φοβάμαι ότι αυτό θα αποδυναμώσει έτσι περαιτέρω την, τις σχέσεις των κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρωτού λοιπόν το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να κοιτάξουμε και το σκέλος των εσόδων. Και εδώ θα διαπιστώσουμε ότι σε διάφορα κράτη-μέλη έχουμε τεράστια προβλήματα σε ό,τι αφορά το σύστημα φορολόγησης. Και υπάρχουν φορολογικά κενά, χάσματα. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε μια εξαιρετική ευκαιρία στην παρούσα φάση. να ενδυναμώσουμε, να ενισχύσουμε το φορολογικό σύστημα προκειμένου να χρειαζόμαστε πιο πολλά, να ε, λαμβάνουμε πιο πολλά έσοδα. Δεν ε, λέω ότι αυτή θα είναι η μαγική λύση που θα λύσει όλα τα προβλήματα, αλλά έχει έρθει πραγματικά η στιγμή να κοιτάξουμε και το θέμα αυτό. Να μην προβαίνουμε διαρκώς και μόνο σε περικοπές. Κυρίε και κύριοι, πολλά κράτη έχουν εδώ πέρα προβλήματα. Δεν είναι δυνατόν. να αποφεύγουμε διάφορα προβλήματα. Δεν μπορούμε, για παράδειγμα, σε θέματα άμυνα να υπολογίζουμε μόνο στο ΝΑΤΟ. Το ίδιο ισχύει και σε ό,τι αφορά τα θέματα γεωργία. Η γεωργία αποτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τα τρόφιμα ή ασφαλή φοδιασμό, αποτελεί σημαντικό σκέλο για την Ευρώπη. Όλα αυτά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριο Ζαν Κλοντ Μικαλεφ από τη Μάλτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από τι διάφορε εισηγήσει που άκουσα εδώ στην Επιτροπή. Έχω να πω το εξή. Η Επιτροπή προφανώ και εξετάζει τα επόμενα δημοσιογενικά μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν και στα θέματα ασφάλειας μεταξύ άλλων. Μου κάνει εντύπωση η έλλειψη. αυτό που με ανησυχεί σε αυτά που άκουσα είναι το εξή. Έχουμε πολλά στοιχεία τα οποία είναι διαφορετικά. Ένα όμως στοιχείο φαίνεται ότι είναι κοινό μεταξύ κρατών μελών. Ένα στοιχείο επί του οποίου συμφωνούν όλοι. Όλοι κοιτάνε τι μπορούν να βγάλουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τι τους αναλογεί, αλλά δεν κοιτάμε ιδιαίτερα το πώς μπορούμε να συνεχίσουμε να φροντίσουμε αυτό το οποίο στην τελική ανάλυση αποτελεί την πηγή των ε, εσόδων αυτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι εφαρμόζει αυτή την ε, λύση, την ενιαία για όλους, μία λύση για όλους. Αυτό δεν μπορεί να είναι αποδεκτό. Χρειαζόμαστε πραγματικούς μηχανισμούς, διαφορετικούς μηχανισμούς, οι οποίοι θα προωθούν τα οικονομικά μέσα, την κοινωνική συνοχή, τα κοινωνικά μέτρα, προκειμένου να μπορέσουν οι χώρες να αναπτυχθούν με έναν ενιαίο, αν και αξιοδομικευμένο τρόπο. Ακολουθώντας δηλαδή τις πολιτικές ε, ευρωπαϊκές, όταν μιλώ για ευρωπαϊκές πολιτικές, το λέω γιατί Φαίνεται ότι παρόλο που όλοι είμαστε τμήματα και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή η ευρωπαϊκή νοοτροπία δεν φαίνεται να μας διέπει όλους. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε έναν προπολογισμό ο οποίος θα καλυπτεί τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Τι νόημα έχει όμως να φροντίσουμε το περιβάλλον και να μην φροντίσουμε την κοινωνική πτυχή και την οικονομία. Όλα αυτά λοιπόν θέλω να πω ότι θα πρέπει να τα κοιτάξουμε από κοινού. Δεν μπορούν να αποτελούν ξεχωριστούς πυλώνες. Γι' αυτό λοιπόν Πιστεύω ότι θα πρέπει να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα και θα πρέπει να δούμε πώς τα δημοσιονομικά μέτρα θα μας επιτρέψουν να ξεπεράσουμε θέματα σε ό,τι αφορά την παρανομή μετανάστευση, θέματα εγκληματικότητας, διακίνηση ανθρώπων. Να κοιτάξουμε επίσης και τον προπολογισμό ως έναν τρόπο να αντιμετωπίσουμε τους μεμονωμένους περιορισμούς που έχει κάθε χώρα. Θα πρέπει τελικά να έχουμε ένα υπολογισμό ο οποίος θα δώσει δύναμη στους πολίτες, όχι σε άλλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Πρόεδρος. Αυτά ήταν τα αιτήματα που λάβαμε για παρεμβάσεις. Ολοκληρώνεται λοιπόν το σημείο αυτό της ημερήσιας της συζήτησης και να δώσω το λόγο στον κύριο Ματελιάν, Πρόεδρο, να κάνει τα καλλιτικά σχόλια. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω κροατικά. Σας ευχαριστώ για την εξαιρετική οργάνωση της Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας και της σημερινή συνεδρίασης. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους αγαπητοί συνάδελφοι για αυτή την επικοδομητική και ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ακούστηκαν κάποια ισχυρά επιχειρήματα, Μερικές φορές ήταν αντικρουόμενες οι θέσεις που εκφράστηκαν. Όμως ε, αυτή η πολυμορφία και η διαχείρισή της ε, είναι ουσιαστικά ένα μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι στο ότι αυτοί οι στόχοι που έχουν εκφραστεί και στην ανακοίνωση της Επιτροπής και στις κατευθυντήριες γραμμές της νέας Επιτροπής αλλά και στις προτάσεις που εκφράστηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ότι αυτοί οι στόχοι έχουν τεθεί πολύ ψηλά και το να τους πετύχουμε, για να τους πετύχουμε θα χρειαστούμε μεγάλες επενδύσεις και προσαρμογές. Όμως βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη συνένεση σε σχέση με τις κοινέ προτεραιότητες από τη σημερινή συζήτηση που ολοκληρώθηκε μόλις, σημειώνουμε ότι δύο θέματα αλλήλω σχετίζονταν. Και αυτό είναι κάτι που αποκάλεσαν κάποιοι παλιές πολιτικές και νέες πολιτικές. Σε ό,τι αφορά στις νέες πολιτικές, μία είναι η Πράσινη Συμφωνία. Καθώς προέρχομαι από την Κροατία, ε, μια χώρα η οποία βασίζεται στο τουρισμό για το 20% του ΑΕΠ της, ε, θέλουμε να επικεντρωθούμε στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βιοπικιλότητα. Γιατί το περιβάλλον και οι άνθρωποι είναι η μεγαλύτερη αξία μας. Η διαχείριση του περιβάλλοντος είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η Κροατία έχει ε, μακρά εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης και Καλωσορίζουμε την ε, ενδυνάμωση της προστασίας των συνόρων και μεγαλύτερο ενεργητικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στη διεθνή βοήθεια. Ακούστηκαν ε, και κάποια σχόλια για πιθανή κρίση που μπορεί να επίκειται. Όμως ε, το να επενδύσουμε περισσότερο στην έρευνα και στην ανάπτυξη και στην καινοτομία, αυτά δεν αφορούν το μέλλον, γιατί χωρίς νέες τεχνολογίες και ψηφιοποίηση δεν μπορεί να υπάρξει βελτίωση της οικονομίας ή οικονομική ανάπτυξη. Ούτε θα υπάρχει ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Τις νέες πολιτικές λοιπόν θα πρέπει να οθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς ένα στόχο που όλοι θέλουμε να πετύχουμε την επόμενη δεκαετία και αυτό να μπορούν να το αναγνωρίσουν οι πολίτες. Όμως επίσης θα πρέπει να γνωρίσουμε ότι αν τα θεμελιά μας δεν είναι ισχυρά, το να οικοδομήσουμε πάνω τους ε, δεν θα φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Σε ό,τι αφορά την ε, σύγκληση μεταξύ των περιοχών, εκεί εφαρμόζονται παραδοσιακές πολιτικές. Ε, τα τελευταία χρόνια οι Κροάτες ε, βλέπουν τα ωφέλη της κοινή αγροτικής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής. Γιατί όταν μιλάμε για πολιτική συνοχή, μιλάμε για ευρωπαϊκά κονδύλια. Και σήμερα τα ευρωπαϊκά κονδύλια είναι ένα από τα πια αναγνωρίσιμα ωφέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα πρέπει να τα εγκαταλείψουμε. Επομένως, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι μετά τον Brexit, αφού αποχώρησε ένα κράτο μέλο, ένα προπολογισμό πρέπει να είναι ευέλικτο και αποτελεσματικό. Επίση, είναι δημοσιονομική περίοδο απαιτεί την επίτευξη της συμφωνίας για τις πολιτικές χρηματοδότησης που συζητήσαμε σήμερα. Όλοι γνωρίζουμε ότι αν δεν θέλουμε κενό στις εκτελεστικές πολιτικές και στα προγράμματα θα πρέπει να δράσουμε υπεύθυνα και να σεβαστούμε τις προθεσμίες. Εγώ ελπίζω ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την Πέμπτη θα δώσει το απαραίτητο έναυσμα. Κάποιοι είπαν ότι χρειάζεται να γίνει θαύμα, αλλά αν συμβεί αυτό η Κροατία, όπως γνωρίζετε, είναι έτοιμη να συνεχίσει στενή και εντατική συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το επόμενο στάδιο της διαδικασίας. Κύριε Πρόεδρε, ήταν τιμή μου να συμπροεδρεύσω μαζί σας αυτή τη συνεδρίαση. Επιτρέψτε μου, αγαπητοί συναδελφοί, να σας δώσω και κάποιες τεχνικές πολιτήριες. Ε, ε, θα ακολουθήσει ένα δείπνο κοκτέιλ που θα ξεκινήσει στις 7 και 4 στον οίκο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Οι κλητήρες περιμένουν ε, μπροστά στην αίθουσα ε, για να σας συνοδεύσουν ε, στον οίκο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας και μην ξεχάσετε τα προσωπικά σας αντικείμενα. Σαν δάσκαλος τα είπα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ολοκληρώνεται εδώ η συνεδρίασή μας.